Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ας ξεκινήσουμε. Έχετε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης μπροστά σας. Έχετε κάποια σχόλια για την ημερήσια διάταξη. Όχι. Άρα προχωρούμε στο επόμενο σημείο, έγκριση των πρακτικών. Αν είστε ικανοποιημένοι, θα προχωρήσουμε από τα κείμενα των πρακτικών, θα προχωρήσουμε στην έγκρισή τους. Συμφωνούμε, βλέπω. Σημείο 3. Ανταλλαγή απόψεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Καταρχάς πρέπει να ζητήσω συγγνώμη δεν είναι πολλοί συνάδελφοι παρόντες. Δεν έχουν συνηθίσει συνάδελφοι στο να ξεκινάμε στην ώρα μας, από ό,τι φαίνεται. Θα το συνηθίσουν όμως. Ο κύριος Μάρσελ Βεσλάιπ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνδρόμων είναι μαζί μας. Θα, κάνει, θα κάνετε την παρουσίασή σας. Θα ξεκινήσουμε και μετά θα ζητώσω το λόγο στους υπόλοιπους. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρήσουμε. Όπως σας είπα, το σφυράκι δεν σας απειλεί, απλά όταν το κουνάω σημαίνει ότι τελειώνει η ώρα σας. Να το θυμάστε. Μπορώ και να το χρησιμοποιήσω, δηλαδή να σας χτυπήσω, αλλά δεν θα το κάνω. Κύριε Βέσλιπ, σας δίνω το λόγο και σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα το απόγευμα για να περάσετε κάποιο χρόνο μαζί σας. Ευχαριστώ. Τιμή μου είναι να είμαι εδώ σήμερα στην Νέα Επιτροπή Μεταφορών, παρότι γνωρίζω κάποια μέλη σας. Μου είπαν ε, ότι έχω 15 λεπτά για να μιλήσω για το ρόλο της υπηρεσίας μου και τις δραστηριότητε. Να σας δώσω και μια χρονολογική προσέγγιση του τι έχουμε κάνει με τα πρώτα πέντε σχεδόν χρόνια της ύπαρξής μας. Το 2005 ξεκίνησαν, ε, ξεκίνησε να λειτουργεί στην ουσία ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ιδιοδρύμων και γρήγορα φάνηκε ότι σε δύο βασικέ οδηγίε ε, στηριζόμαστε την ασφάλεια και την διαλειτουργικότητα. Εξ αρχή ε, θέλαμε να δούμε το πρόγραμμα στο σύστημα, στον τομέα των ATR και μα ζητήθηκε να λειτουργήσουμε σαν αρχή συστήματος με το, το ERTMS, την εξέλιξη ERTMS και μια... δημιουργήσαμε μια, γρήγορα μια ομάδα, μονάδα αξιολόγηση για να κρίνει τις προτάσεις και συστάσεις της υπηρεσίας του, του οργανισμού. Καταρχάς, η πρώτη μας συνάντηση ήταν με τις Εθνικές Αρχές Ασφάλειας το Σεπτέμβριο, την 1η Σεπτεμβρίου του 5 είναι πολύ σημαντικό να σας θυμίζω ότι οι εθνικές αρχές, και πάλι αυτό αποτελεί εξαίρεση στον συνδρομικό τομέα, δημιουργήθηκαν παράλληλα με την, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, με κάποιες διαφορές βέβαια από κράτος σε κράτος. Παράλληλα, ξεκινήσαμε με την πρόσληψη ειδικών για τη δημιουργία μιας λευκής βίβλου με στόχο να έχουμε άτομα με προσόντα και με γνώσεις στον τομέα, στον οργανισμό μας. Ένα άλλο θετικό είναι ότι ο κλάδος εξ αρχής ε, έδειξε εσφουσιώδη υποστήριξη σε αυτά που κάνουν, επικρίνοντας τα ενδεχομένως, ε, αλλά έστειλαν στον οργανισμό ειδικού με, πολύ καλέ με πολύ καλές γνώσεις σε διάφορους τομείς του κλάδου. Το 2006 ξεκινήσαμε από την πρώτη πρώτη του 2006 να αναπτύσσουμε το σύστημα το ERTMS System Management. Πρώτη χρονιά ήταν πραγματικών εξελίξεων σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες που, είχαμε, που είχαν τεθεί με τον ιδρυτικό κανονισμό και είχαμε τη δυνατότητα να υιοθετήσουμε το EAIF, μια οργάνωση του κλάδο που κάλυ, πήραμε όλε τι δραστηριότητε του οργανισμού αυτού. Ασχολιόντουσαν κυρίω με διαλειτουργικότητα, υψηλέ ταχύτητε κλπ. Επίση, ήμασταν ο πρώτο οργανισμό που υπόγραψε ένα μνημόνιο συνεννόηση με την Επιτροπή για να ορίσει εξ αρχή τι διαφορετικέ ευθύνε, ε, τα καθήκοντα και του ρόλου των δύο πλευρών. Ήταν κάτι πολύ χρήσιμο, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε, αλλά το παράδειγμα αυτό έκτοτε το ακολούθησαν άλλοι τρει οργανισμοί ξεκινήσαμε να δουλεύουμε για τις ε, τεχνικές προδιαγραφές παραδοσιακών σιδηροδρομών. Από το ξεκίνημα ε, του έτους ε, βάλαμε, δημιουργήσαμε τον πίνακα ελέγχου του ΙΑΤΜΣ και την συμβουλευτική ομάδα. Ε, να σας πω, για να μην είναι πολύ θεωρητική συζήτηση, από το προβλήμα του, του είναι ότι υπάρχουν πάνω από 100 αιτήματα έχουν υποβληθεί το 2005. Εμείς θελήσαμε να κάνουμε να περάσουμε μέσω, αναγνωρισμένων, μέσω αναγνωρισμένων ε, οργανισμών και ο αριθμό των εδημάτων περιορίστηκε τελικά κατά 60% τους πρώτους δύο μήνες. Συνεργαστήκαμε επίσης και με τις οργανώσεις ε, κοινοποιήσει και με τη Σενσιμινέκ και την έτσι τις ε, συνδικαλιστική οργανώσεις. Επίση, δημιουργήσαμε μια σειρά υποδομών, πήρατε σχετικέ πληροφορίε και αναπτύξαμε και το πρώτο σύστημα τεχνολογία πληροφόρηση και επικοινωνιών του οργανισμού. Δημιουργήσαμε μια διαχειριστική επιτροπή με τρεις με, τρία μέλη τη είναι παρόντα εδώ σήμερα και έχουμε στόχο να ξεκαθαρίσουμε τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων πλευρών του, της υπηρεσίας. Το 2007 παρουσιάσαμε το πρώτο συμβατικό TSI Infrastructure, το πρώτο, CMS, το πρώτο CMS, το την ενδιάμεση έκθεση για τα οχήματα ε, για τα χήματα επιβατών και του δρόμους και επιπλέον είχαμε και τον ορισμό της μελλοντική ενίσχυσης της τρίτης version της τρίτης εκδοχής του ETCMS. Επίσης ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με τους συντονιστές των διαδρόμων, το μήνυμα του ρόλου μας είναι αυτό. Θέλουμε να προσφέρουμε συνεργασία και να βοηθήσουμε τις δομές αυτές σε μια σειρά διαστηριοτήτων, οικονομική αξιολόγηση, ATMS, ε διαλειτουργικότητα. Συνεργαστήκαμε με την OTIF, τους επόμενους μήνες θα ακούσετε πολλά για την OTIF και την OSJD, τον Παλιό Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Σοβιετικής Ένωσης. Επίσης έχουμε δημιουργήσει μία από τα δύσκολα και περίπλοκα ε, τη δύσκολη και περίπλοκη διοικητική διαχείριση των ε, δομών. Το 2007 έγινε σαφές ότι ο ρόλος του οργανισμού έπρεπε να εξελιχθεί ταχύτερα. Όπως αυτή τη στιγμή θα ακούσετε στην γλώσσα μας να μιλάμε για open points, ανοιχτά σημεία. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι σημεία που έχουν συζητηθεί επί δεκαετίες μερικές φορές χωρίς λύση. Έχουμε λοιπόν μια πρόσφατη εντολή να κλείσουμε όλα τα ανοιχτά σημεία, τα ανοιχτά θέματα στο TSI και σε άλλα κείμενα. Κάτι πολύ φιλόδοξο. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε τις συζητήσεις και για το νέο νομικό πλαίσιο του οργανισμού που τοποποιήθηκε τελείως ε, πέρσι, στο τέλος του περσινού έτους. Αυτό εξ αρχής έδειξε ότι υπάρχει μια πραγματική βούληση όλων των πλευρών του κλάδου να ενισχύσουν την εμβέλεια και το πεδίο και τον χώρο των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Επίσης οργανώσαμε μια πολύ σημαντική συζήτηση με την NSA, θα επανέλθω στο θέμα αυτό, τις Εθνικές ε, Αρχές Ασφάλειας δηλαδή και ξεκινήσαμε να προχωρούμε στην πρώτη, στα πρώτα βήματα της ε, ε, προσέγγι, των προσεγγίσεων με τα peer reviews. Το 2008 ξαναρχίσαμε να λαμβάνουμε υπόψη τις απαιτήσει που προκύπτουν από την συνδιαλλαγή που προέκυψε για το τρίτο συνδρομικό πακέτο και από ό,τι φαίνεται ε, τα, τα, ίδια συμπεράσματα φτάνουν ε, και οι συμβαστικές ε, προτάσεις. Επίσης προβλέφθηκε να έχουμε το συντομότερο δυνατό δραστηριότητε για τις ε, τι αμοιβέ αποδοχέ. Θα σα αναφέρω και κάτι άλλο, ο συνάδελφο Πατρίκ Κουντού από την υπηρεσία, από την ε, υπηρεσία αεροπορικών μεταφορών ε, καταγγέλθηκε από τον κύριο Γκαλουάδη ότι αυτό ε, κόστισε περίπου ένα εκατομμύριο και μας είπαν ότι ο κύριος Γκαλουά δήλωσε ότι ε, για ένα αεροσκάφος το κόστος ήταν πολύ μεγαλύτερο από ότι για ένα ε, για μια σιδηροδρομική μηχανή και άρα ο κλάδος ε, χρειάζεται να αναπτύξει την αμοιβαία αποδοχή. Αυτή τη στιγμή αποφασίσαμε δείχνοντας ελληνική στην, στον οργανισμό να ξεκινήσουμε εκ των προτέρων τη δραστηριότητα αυτή με τη διαδικασία, με τη δημιουργία της μονάδας αμοιβαίας αποδοχής. Επίσης, ε, ε δεχθήκαμε την τέταρτη εκδοχή του ETMS, το 2,3 OD, και χαίρο που δεν μιλάμε πολύ για το ETMS, γιατί από ό,τι φαίνεται λειτουργεί μια χαρά. Επίσης, είμαστε μέσα στο χρονικό πλαίσιο να ξεκινήσουμε τον διαγωνισμό για, την, ε, για να βγει εμπορικά το baseline 3 πριν το τελειώσει το έτος. Όπως σας είπα, δουλέψαμε και με νέες πρωτοβουλίες, την αμοιβαία αποδοχή, την έγκριση τύπου, την πιστοποίηση ε, ENTT, κάτι πολύ σημαντικό, και γρήγορα φάνηκε ότι με τις νέες οδηγίες, τον νέο κανονισμό, τις νέες εντολές, τις νέες εμπλοκές ε, των ε, διαφόρων πλευρών, η αύξηση των ετοιμάτων δημιούργησε πίεση στον οργανισμό. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε στην Επιτροπή το πρόγραμμα εργασία για το 2010 και τον προπολογισμό και το πρόγραμμα εγκατάσταση. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, με, να δουλέψουμε σε ένα σταθερό νομικό περιβάλλον. Είναι ουσιαστικό αυτό για να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη δραστηριοποίηση όπως αυτή που απαιτείται στον τομέα των σιδηροδρόμων. Επίσης, ε, ενσωματώνουμε την ε, χρησιμοποίηση εμπειρία σε νέε τεχνολογίε στην ανάπτυξη νέων κανόνων και όλο και περισσότερο συνεργαζόμαστε με τι διάφορε πλευρέ. Πάντα επαναλαμβάνουμε ότι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων είναι το μόνο σημείο στην Ευρώπη όπου συναντούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο. Και ξέρετε ότι στον κλάδο των σιδηροδρόμων υπάρχουν πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι. Ε, εθνικέ Αρχέ Ασφάλεια, εννέα αναγνωρισμένοι οργανισμοί, ε, η NB Rail, ε, πάρα πολλέ εθνικέ. Είναι πλεονέκτημα αυτό, αλλά κάθε φορά που εμφανίζεται ένα ζήτημα συντονισμού και συνοχής, στρέφονται όλοι σε εμά. έχετε ένα, μια σειρά διαφανειών που βλέπετε πώς δουλεύουμε. Δουλεύουμε με τους αναγνωρισμένους ε, πιστοποιημένους τομείς του κλάδου, CER, AIM, EAFA, UITP, δημόσιες μεταφορές UIIR, συνδυασμένες μεταφορές, UIP, UNIFE, τον κλάδο και την ETF. Η e ETF είναι ε, η Ένωση των Συνδικάτων. Αυτές είναι οι πρώτες κατηγορίες εταίρων του οργανισμού μας. Μετά έχουμε ειδικού από τις 26 εθνικές αρχές ασφάλειας και η Νορβηγία, παρεπιπτόντως και να σας πω, μετέχει στις δραστηριότητε μας και δραστήρια και όλες. Είμαστε Έχουμε την προεδρία των ομάδων εργασία του οργανισμού με την οριζόντια υποστήριξη τη ομάδα οικονομικού ελέγχου, οικονομική παρακολούθηση. Παρέχουμε συστάσει. Η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον συνένεση. Εμείς ε, αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Ο διευθυντής αναλαμβάνει την τελική ε, ευθύνη για τις συστάσεις. κατόπιν μετά από διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους ε, των πελατών τόσο επιβατών όσο και εμπορευματικών μεταφορών ε, πηγαίνει στην Επιτροπή Κινδύνου αύριο θα συναντηθεί εδώ στις Βεξέλλες είναι Επιτροπή των Κρατών Μελών και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατόπιν η παραδοσιακή δομή είναι η διαφορά είναι η ο μεγάλος αριθμός των εκπροσώπων και εταίρων. Να συνεχίσω στα γαλλικά. Θέλω στο μικρό χρονικό διάστημα που έχω, γιατί κυρίω θέλω να απαντήσω ερωτήσει. Θα προσπαθήσω συμπερασματικά να συνοψίσω συμπερασματικά τις προκλήσεις του οργανισμού του επόμενου έτη. Σε δύο-τρία χρόνια πρέπει να Αυτό εδώ βλέπετε όλη την συνδρομική δομή που πρέπει να συμπληρώσουμε. Τωρινέ τεχνικές προδιαγραφέ για το ευρωπαϊκό, διευρωπαϊκό δίκτυο και το τροχαίο υλικό. Θα πρέπει να επεκτείνουμε τον τομέα των STI για να καλύψουμε όλα τα δίκτυα. Να δούμε ας πούμε πού σταματά το τοπικό αστικό περιφερειακό δίκτυο και πού αρχίζει το συνδεδομικό. Το cross section είναι το, το cross acceptance ε, άλλαξε τη φιλοσοφία του οργανισμού. Θα καθορίσουμε τους κανόνες για το μέλλον για να καθορίσουμε και τις επενδύσεις, ενώ τώρα στην cross acceptance θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την υφιστάμενη κατάσταση, να εξετάσουμε τους εθνικούς κανόνες, να ορίσουμε τις ισοδυναμίες και να καταλήξουμε στο να μην χρειάζεται να γίνεται 25 φορές έλεγχος της ίδιας μηχανής από ε, παρόμοιους ε, τεχνικούς. Το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας ισχύει για τις ε, συνδρομικές επιχειρήσεις. Είναι ένα σύστημα κλασικό αυτό. Πιστεύουμε ότι θα τελειώσουμε σε 2-3 χρόνια τις βασικές δουλειές για τα STI, για τις μεθόδους ασφάλειας. Όλο και περισσότερο χρειάζεται να εξηγήσουμε ε, θέματα συντήρησης, ε, πλοήγησης και συνδρομής, να περάσουμε το 2012 τη νέα εκδοχή του ERTMS e, e και να, κάτι πολύ σημαντικό, αναπτύξουμε τον ρόλο της αμοιβαίας αναγνώρισης κανόνων, συστημάτων και διαδικασιών μεταξύ κρατών μελών, εθνικών αρχών και εμπλεκομένων φορέων. Αυτό το μνίζει εκ το βασικό ρόλο των εθνικών αρχών. Στον τομέα των αερομεταφορών υπάρχει βασική ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, γιατί οι οργανισμοί δεν υπάρχουν. Εμεί, ωστόσο, δημιουργηθήκαμε ταυτόχρονα με τι εθνικέ αρχέ, με κάποιε εξαιρέσει στη Γερμανία, στη Βρετανία, αλλά είναι εξαιρέσει. Σήμερα οι διάφορε εθνικέ αρχέ ασφάλεια έχουν ε, προσωπικό από 10 μέχρι 1.300 άτομα. Μέσο όρο είναι 100. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε δεν έχουν τις, ευθύνες, τις δυνατότητες που μπορούν να έχουν, ενώ έχουν τεράστιες ευθύνες. Δίνουμε λοιπόν πάρα πολύ χρόνο και μέσα στη συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Στην διάσκεψη που έγινε μετά το ατύχημα στο Βιαρέτζιο, ο αντιπρόεδρος κ. Σταγιάννη αναφέρθηκε σε πέντε βασικά ζητήματα την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου και των εξουσιών του οργανισμού. και έστειλαν, ο κλάδος έστειλε και μια σχετική επιστολή στον Αντιπρόεδρο ζητώντας την ενίσχυση του ρόλου του, του οργανισμού. Ε, βέβαια, ε, αυτό έχει και μερικέ αντιφάσει. Κάποιοι ειδικοί λένε ότι δεν προλαβαίνουν να παρακολουθήσουν το ρυθμό δουλειά μα. Κάποιες ελληνικέ αρχές ζητούν να περιορίσουμε την ταχύτητα των δραστηριοτήτων μας και Επιπλέον χρειάζεται να ολοκληρώσουμε και τη λειτουργία του οργανισμού. Είναι σημαντικό, είναι προφανές, α, κάτι που ξέχασε και ξεχνάμε συχνά και εξηγεί ακριβώ την σημασία της δράσης του κλάδου είναι ότι ο σιδηροδρομικός τομέας είναι δυστυχώς ένας από τους τελευταίους κλάδους όπου είμαστε στην πρωτοπόρη στην Ευρώπη, 72% των εμπορευματικών μεταφορών στον κόσμο. Είναι λοιπόν σημαντικότατο να αναπτύσσουμε ευρωπαϊκούς κανόνες επαρκώς ισχυρούς για να υιοθετηθούν παντού. Στα πλαίσια, σε ό,τι αφορά το ETMS, αφού βάλαμε κάποια τάξη στην ανάπτυξη του ETMS, είδατε ότι αμέσως υιοθετήθηκε από την Αυστραλία, το Μεξικό, το, το δοκιμάζουν στην Κίνα και την Ινδία, υιοθετήθηκε από την Σαουδική Αραβία και το Μαρόκο. Οι τελευταίες χώρες που το υιοθέτησαν ήταν Νέα Ισλανδία και η Λιβύα. Προφανώς αυτό δεν το χρησιμοποιούν για να υπάρχει διαλειτουργικότητα με το ευρωπαϊκό σύστημα, αλλά γιατί είναι ένα σύστημα εύκολο, ε, προσπελάσιμο και το οποίο που βγαίνει στην αγορά. Επίσης, δημιουργήσαμε με τις εθνικές αρχές μια ομάδα περισυλλογής, διότι είναι σαφές και η συζήτηση αυτή έχει γίνει ήδη στο παρελθόν στο, στην Επιτροπή σας να αναφέρω, ότι η ενίσχυση της συνεργασίας και του ελέγχου, του auditing και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εθνικών αρχών είναι κάτι το ιδιαίτερα αναγκαίο και θα είναι και κρίσιμο στιγμή για την ανάπτυξη του συστήματος. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια ομάδα περισυλλογή με τι εθνικέ αρχές, δεν υπάρχει λοιπόν σύγκρουση αρμοδιοτήτων, που θέλει να εξετάσει το πώ θα εξασφαλιστεί μια ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών. Αυτή ήταν μια σύντομη παρουσίαση. Ελπίζω ωστόσο ότι πήρατε όλοι αυτό το USB stick που έχει όλα τα στοιχεία και τα διάφορα κείμενα. Πρόκειται για ένα παράδειγμα της εξέλιξης της ασφάλειας στην Ευρώπη. Το 1970 υπήρχαν περίπου 400 ειδικού στα 15 τότε κράτη-μέλη της Ένωσης. Σήμερα είναι 100. Λιγότερο από 100, καμία 40 υπολογίστηκαν στα 25 κράτη-μέλη. Ε, εμείς λοιπόν δεν είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε την ασφάλεια των σιδεδομών αλλά κρατήσουμε την υψηλή την εξαιρετικά υψηλή επίδοση των σιδεδόμων στην αγορά μας. Κάτι τελείως διαφορετικό με άλλες χώρες που έχουν απελευθερώσει το σύνολο, το σύστημά τους. Η εξέλιξη είναι ίδια, τα ίδια τα βλέπετε στην έκθεσή μας και πολύ καλύτερα μάλιστα. Ξέρουμε λοιπόν ότι πολλές νέες δραστηριότητε θα αναλυθούν από την υπηρεσία μας. Το ίδιο ίσχυσε τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι μόνιμα μια πρόκληση, και φορά φαίνονται δύσκολα τα πράγματα. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πιστεύουμε ότι η επόμενη εξέλιξη θα είναι ενίσχυση της αμοιβαίας εντυπο... Ε, εμπιστοσύνη μεταξύ των αρμόδιων εθνικών φορέων και ισχυρότερος ρόλος για τη δική μας υπηρεσία. Αυτά και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Um, ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Οι συντονιστές θα ξεκινήσουν τη συζήτηση. Ένα τρίλεπτο ο καθένας. Κύριος Γκρό για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Θα είμαι πολύ σύντομο όσον αφορά την ερώτησή μου. Απαντήσατε εν μέρη στο ερώτημά μου. Είπατε ότι έχουμε πρόκληση για το μέλλον. Πώς βλέπετε την υπηρεσία που θα μπορεί να αντικαταστήσει με την πάρο των ετών τις εθνικές αρχές. Πώς το βλέπετε αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο. Κάτι που αφορά περισσότερο την ασφάλεια και τη φιλελευθεροποίηση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Απαντήσατε μέρη σε αυτό. Πώς βλέπετε μεσοπρόθεσμα την εγγύηση ασφάλειας στο δίκτυο εν γέννη, προχωρώντας ταυτόχρονα στην ε, φιλελευθεροποίηση της αγοράς. Και τρίτον, διαλειτουργικότητα, τεχνική διαλειτουργικότητα. Κατά την άποψή σας, πώς εκτιμάτε τις προσπάθειες, τις σημαντικότητες που πρέπει να γίνουν όσον αφορά την τεχνική διαλειτουργικότητα. Δοθέντως ότι γνωρίζω ότι είναι ένα από τα δεινά από τα οποία υποφέρει περισσότερο ο σιδηρόδρομος, οι σιδηρομικές μεταφορές, από ότι όλες οι άλλες μεταφορές στην Ευρώπη, τα λέει μεταφορά. Ευχαριστώ. Ο κ. Ελκ Ρόγια, του Κύριος Μάκενροε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας που μας κάνατε για την υπηρεσία. Είναι μια υπηρεσία που ακόμα οικοδομείται. Αυτό είναι ξεκάθαρο, προχωρήσατε πολύ, αλλά απομένουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Αναφερθήκατε σε διάφορα θέματα. Είναι δύσκολο, πιστεύω, να διαχωριστεί η υπηρεσία σας από τα τεκτενόμενα στο σιδηροδρομικό τομέα. Εκεί έχουν εμφανιστεί τεράστιες προκλήσεις. Τις πρόσφατες εβδομάδες είχαμε άσχημες ειδήσει. Για τη μεταφορά αγαθών τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα, για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο και, άλλα, και ένα άλλο κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει προβλήματα σε αυτό το τομέα. Πολλοί παράγοντε παίζουν ρόλο σε αυτό. Η οικονομική συγκυρία καταρχά, αλλά και άλλοι παράγοντε. Ο ίδιο αναφερθήκατε στην ανάγκη για κοινέ προδιαγραφές ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά με το σωστό τρόπο, ότι χρειάζονται επενδύσεις, είναι το θέμα της αξιοπιστίας, της ακρίβειας των σιδεοδρόμων, των δρομολογίων της ακρίβειας. Για την υπηρεσία σας τώρα. Πιστεύετε ότι μπορεί να παίξετε ένα ρόλο βοηθώντας να πετύχουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται να τις συντονίσετε τις μεταρρυθμίσεις. Ποια είναι τα σημαντικότερα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ούτω ώστε οι σιδηρόδρομοι να αποκτήσουν ξανά το μερίδιο της αγοράς που είχαν. Ακούω ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού μεταξύ επιχειρήσεων διαχείρισης υποδομών είναι πρόβλημα για να λειτουργούν σωστά οι διεθνείς μεταφορές και οι διασυνδέσεις. Δεν ξέρω αν η υπηρεσία σου μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Και τέλο, όπως είπε ο κύριος Γκρός, πώς βλέπετε την, ε, στην υπηρεσία σας. Χρειάζεται περισσότερες εξουσίες, ποιες και αν ναι, πότε πιστεύετε ότι θα έρθουν. Ο κ. Κράμερ για τους πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας. Έχω να κάνω τέσσερις ερωτήσεις. Πρώτον, υπάρχουν ήδη συγκρούσεις με την cross acceptance, την αμοιβαία αποδοχή, όπου κάποιες χώρες λένε ότι εμείς δεν δεχόμεθα αυτό το σύρμο ή μήπως δεν έχετε εμπειρία από αυτού. Είναι ίσως πολύ νωρίς. Δεύτερον, για το ATMS λέτε ότι μοιάζει να λειτουργεί πολύ καλά και ερωτώ, είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρχει συγχρηματοδότηση εάν το RTMS ε ε, επεκταθεί. Ξέρετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ανάμεσα στο Βερολίνο και το Ρόστοκ. Αυτό ε, λύθηκε και υπάρχουν άλλες παρεμφερείς συγκρούσεις όπως τη ERTMS κατόπιν. Όσον αφορά τον φορέα σας. Έχετε κάποια νομική βάση, πρέπει να επεκταθούν ενδεχομένως οι αρμοδιότητές σας ή μήπως ε, είσαστε ικανοποιημένοι και απλά χρειαζόσαστε περισσότερα χρήματα και περισσότερους εργαζομένους. Και με, κατόπιν, τι γίνεται με το περιβάλλον. Γνωρίζουμε ότι η ΕΑΖΑ έχει συστήσει ένα κέντρο αρμοδιοτήτων. Ε, βεβαίως ε, και οι σιδηρόδρομοι είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, όμως προκαλούν θόρυβο, καταναλώνουν ενέργεια και το το πρόβλημα είναι η διαλειτουργικότητα. Εσείς έχετε κατά νου να συστήσετε κάτι τέτοιο έχοντας κατά νου και το περιβάλλον. Οι σιδηρόδρομοι καταναλώνουν το 25% ε, της ενέργειας και μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και με την ηχορύπανση. Αν λοιπόν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα θα υπάρξει πρόβλημα με το κύρος των σιδηροδρόμων. Έχετε κάποιο πρόγραμμα για το πώς θα αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ ο Αντιπρόεδρος Βαντάλεν ο τελευταίος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εξετάσουμε σημαντικό θέμα, το θέμα της ασφάλειας. Είπατε το σύστημα για την ώρα λειτουργεί, το ERTMS. Θα ήθελα να ξέρω αν πράγματι αυτό συμβαίνει. Στην Ολλανδία τα τελευταία χρόνια Είχαμε σοβαρά προβλήματα με τη μεταφορά εμπορευμάτων σιδηροδρομικά. Στην Πάντρεχ την περασμένη εβδομάδα είχαμε σοβαρά τύχημα. Και διάφοροι φορείς είπαν ότι απέχουμε πολύ από τον ε, επιθυμητό στόχο. Θα έπρεπε να πάμε στο ATB Plus και σύντομα θα δούμε ότι θα έχουμε ένα σύστημα που, ασφαλείας που λειτουργεί στις πολύ χαμηλές ταχύτητες. Για την ώρα δεν προστατεύονται παρκός τα τρένα που κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Κάποιοι φορείς διατείνονται ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα διάμεσο μέσο, ε, βήμα. Στο ATS, το αυτόματο σύστημα ασφαλείας για τα τρένα. Για την επόμενη δεκαετία θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί στι διαβάσει τουλάχιστον για τα τρένα που κινούνται σε χαμηλέ ταχύτητε. Γιατί είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Ποιοι έχουν δίκιο, οι ATS, αυτοί που υποστηρίζουν τα ATS ή το ETRM. Μετά, συζητήθηκε στο, το δυστύχημα στην Barendrecht και συζητήθηκε το θέμα της μεταφοράς εμπορευμάτων, κυρίως στην χώρα μου, διότι εκείνοι που υπερασπίζονται τους σιδηροδρόμους και διοργάνωσαν τη συνάντηση, είπαν ότι πρέπει να λύσετε τα προβλήματα, αλλιώς σας προειδοποιούμε. Θα γίνει ο χαμός μετά την 1η Ιανουαρίου. Υπάρχουν προβλήματα με τα βαγόνια, σπάνιοι άξονες τους και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για την ασφάλεια, τόσο σοβαρά που καθόρισαν προθεσμία οι υπερασπιστές των σιδηροδρόμων. Μέχρι 1η Ιανουαρίου πρέπει όλα να τα έχουμε ρυθμίσει. Διαφορετικά λένε θα σταματήσουμε να μεταφέρουμε εμπορεύματα σιδηροδρομικά. Και έτσι έρχομαι στο τρίτο θέμα μου. Η ασφάλεια στους σιδηροδρόμους. Είναι καλή ασφάλεια, ανησυχώ. Κυρίως μετά το ατύχημα στο Μπάρεντρεχτ, με αυτά που άκουσα με τις επόμενες εβδομάδες, δεν θέλω να ξέρω τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό. Και, και εσείς τι πιστεύετε για αυτό το δυστύχημα. Τι μάθατε για το ατύχημα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Βαντάλε. Κύριε Βασιλάκη. Θες να Θέλετε να απαντήσετε στους πρώτους τέσσερις που έθεσαν τις ερωτήσεις και μετά περνάμε στο δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μαδοποιήσω τις απαντήσεις για να δώσω λεπτομερείς απαντήσεις. Κύριε Γκρός, το πρώτο ερώτημα είναι πολύ ευαίσθητο. Το δεύτερο συνδρομικό πακέτο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, προβλέπει, αυτοιμηθήκαμε, η υπηρεσία για τους υδρόμους ευρωπαϊκούς και εθνικές αρχές για τους γιατί ένας από τους λόγους είναι πώς να το πω τώρα. Τα κράτη-μέλη ήθελαν να έχουν την εποπτεία στα συνδρομικά τους ε, συστήματα. Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο. Επίσης, για να γίνει σωστά ο έλεγχος σε συνδρομικό δίκτυο χρειάζεται πάρα πολύ ισχυρή εθνική παρουσία. Σήμερα, όσοι έχουν οι νόμοι, υπάρχουν ε, κάποιες Έχουμε ρόλο συντονιστικό, λειτουργεί καλά, υπάρχει μεγάλη ζήτηση συντονισμό και όπως είπα πιστεύω ότι εν πάση περιπτώσει επιβάλλει λογική να κινηθούμε προς σημαντικότερο ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο και εποπτεία των δραστηριοτήτων των διαφόρων υπηρεσιών. Γιατί? Διότι εθνικοί φορείς εξορισμού συνδέονται άμεσα με τις μεγάλες ιεροδρομικές επιχειρήσεις της χώρας και τα Υπουργεία και πολύ συχνά στρέφονται προς εμάς διότι η ανεξαρτησία τους θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δυσκολία. Νομίζω ότι αν θα υπάρξει εξέλιξη, πως τα εκεί θα κινηθεί σήμερα κάποιοι συνάδελφοι των εθνικών φορέων. Διστάζουν πολύ, φοβούνται ότι μπορεί να καταργηθούν οι υπηρεσίες τους. Αλλά χρειάζεται μεγάλο συντονισμό. Αυτό είναι θέμα πολιτικό βέβαια να υπερισχύει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία επί των Εθνικών Υπηρεσιών και η δημιουργία του σωστού συστήματο είναι σημαντικά θέματα. Τώρα φιλελευθερωποίηση και ασφάλεια ε, ίσως είναι μια εν μέρη απάντηση αυτή που έδωσα ήδη. Λοιπόν, η ασφάλεια στο συνδρομικό τομέα έχει προτεραιότητα. Το βλέπετε στι όλε αναλύσει που κάνουμε το στάτ, ότι η κατάσταση βελτιώνεται σημαντικά. Έχει βελτιωθεί και η ασφάλεια των σιδηροδρόμων είναι πολύ ανώτερη από όλε τι άλλε άλλα είδη μεταφορών. Όμως, εκτροχιασμοί, ε, ε, θράψεις αξώνων κλπ. συμβαίνουν καθημερινά. Γίνεται σημαντική δουλειά από τη μονάδα ασφάλειας που κάνει ανάλυση, ε, παρακολούθηση, ανταλλαγή εμπειριών κλπ. Όσον αναφέρεστε στα εμπορικά, στις εμπορικές αμαξοστοιχίες, αν πρέπει να σταματήσουν, τότε όλοι θα χρησιμοποιήσουν οδικέ μεταφορέ. Και οι κίνδυνοι με τι οδικέ μεταφορέ είναι πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι με τι δρομικέ μεταφορέ. Το ότι υπάρχει ο κίνδυνο για κάποια ατυχήματα, ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό ο κίνδυνο να συμβούν αυτά τα ατυχήματα, αλλά πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται μακροπρόθεσμα, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα και τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε για να κάνουμε κάτι για αυτά τα προβλήματα. Σα διαβεβαιώ λοιπόν ότι η Task Force παρακολουθεί, εξετάζει το ατύχημα και έχουμε de facto αναλάβει την εφαρμογή του προγράμματο δράση, που δεν έχουμε νομική βάση, ακόμα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα επεισόδια και τα ατυχήματα. Είναι λογικό να υπάρχει ευαισθησία για κάποια είδη ατυχημάτων, αλλά να πάρω παράδειγμα τη φιλελευθερωποίηση στη Βρετανία και αλλού έγιναν δύο-τρία ατυχημάτα. Αν δείτε όμω μακροπρόθεσμα τι εξελίξει του διαδρόμου, σήμερα η Μεγάλη Βρετανία είναι από τι χώρε που είναι στην καλύτερη δυνατή θέση και μισέ προτάσει για θέματα ασφαλεία έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, ποιο είναι το σημαντικό μέσο τη διαφάνεια που θα εφαρμόσουμε. Βλέπετε όλα δημοσιεύονται, τα πιστοποιητικά ασφαλεία και όλα αυτά. Εφαρμόζουμε τη διαφάνεια και την ανάγκη να εποπτεύουμε όλε τι δρομικέ επιχειρήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικός ρόλος που μπορούμε να διαδραματίσουμε στον τομέα. Η διαλειτουργικότητα, η τεχνική διαλειτουργικότητα, τεράστιο θέμα. Ξεκινήσαμε το 1996 με τα τρένα υψηλής ταχύτητας. Τώρα ολοκληρώνεται ο συμβατικός τομέας. Έχει παραγγελθεί νέο υλικό και το υλικό αυτό θα πρέπει να πληρεί τις πιο υψηλέ κοινέ προδιαγραφές για το ευρωπαϊκό σύστημα. Ένα παράδειγμα, θα ακούσατε να αναφέρεται η πιστοποίηση τύπου στον τομέα των αερομεταφορών που καλύπτει διάφορα είδη αεροσκαφών. Ο μέσο μέγεθος είναι 7 ε, 7 ατομικάνες στα πιστοποιητικά τύπου. Και προσπαθούμε να λάβουμε όλα τα τεχνικά μέτρα με την υποστήριξη του τομέα και της βιομηχανίας για να επαφαρμόσουμε τα σωστά μέτρα όσον αφορά αυτήν την κάλυψη. Όσον αφορά ποιες είναι οι δυνατότητες... Ε, για την ώρα τουλάχιστον λοιπόν υπάρχει μια αύξηση στη μεταφορά των επιβατών και Άλλο σημαντικό θέμα και σημαντικό βήμα είναι και ότι χρειαζόμαστε βελτίωση των βαγονιών για τους επιβάτες και γενικά του υλικού. Άλλο πρόβλημα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είμαστε από τους τελευταίους τομείς όπου η Ευρώπη ηγείται στην παγκόσμια αγορά, στο τομέα μας, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι αν θέλεις να στρώσεις 200 χιλιόμετρα νέων σιδηροτροχιών στην Ευρώπη, δεν θα παραγγέλλονται όλες οι τροχές στην, ε, στην Ευρώπη. Κοιτάξτε τι γίνεται στη ΣΥΠΑ, Σοδική Αραβία στην, ε, και αλλού. Θα σταματήσουν οι επενδύσεις σε αερομεταφορές εκεί και θα δώσουν όλα τα χρήματα για τις συνδρομικές μεταφορές στο μέλλον. διαπιστώνεται ότι προχωρούν πιο γρήγορα οι εξελίξεις σε όλο τον κόσμο όσον αφορά τους σιδηροδρόμους. Για τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμων υπάρχουν πραχυπρόθεσμα ευκαιρίες, υπάρχουν προβλήματα βέβαια όσον αφορά την αξιοπιστία και κάποια ποιοτικά προβλήματα, όμως όπως είπε και ο κ. Κράμερ, υπάρχουν προβλήματα και με τις υποδομές. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αν θέλουμε να λάβουμε μέτρα, αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε νέα, νέο εξοπλισμό, πρέπει να σεβόμαστε τις προδιαγραφές που υπόκειται συνεχώς η οικονομική αξιολόγηση. Έτσι, θα κατασκευάζουμε βαγόνια που είναι πιο φθηνά δεν θέλουμε να κοστίζουν οι ετομηχανέ πάρα πολύ ακριβά, πιο ακριβά από ό,τι θα μπορούσαν να κοστίζουν. Θέλουμε να κρατάμε το κόστο χαμηλά. Πρέπει να ακολουθήσουμε τη σωστή προσέγγιση για να βρούμε τις σωστές λύσεις. Είναι επίσης σαφές ότι η εμπιστοσύνη έχει σημασία. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτά που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από πλευρά αρχών. Όταν ελεγχθεί μια ατομηχανή σε ένα ε, κράτο μέλο ή με αμαξοστοιχεία δεν χρειάζεται να ελεγχθεί και από τα άλλα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό απαιτεί εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών. Ότι η έλεγχη που διεξάγει ένα άλλο κράτο μέλο είναι αρκετή και ικανοποιούν το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση στην Ολλανδία. έχει σύστημα RTMS. Αυτό αναπτύχθηκε παράλληλα με το 30D. Παράλληλα δύο συστήματα. Δεν θέλουμε να ξαναγίνει αυτό με την baseline 3 διότι θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται το σύστημα σε όλες τις χώρες και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που επί 10 χρόνια, 11 χρόνια αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τη θέσπιση προδιαγραφών. Στην, στην Ολλανδία υπήρξαν τρία προγράμματα RTMS. Υπήρχαν προβλήματα συντονισμού και υπήρχαν και διαφορές μεταξύ των προδιαγραφών. Δεν θέλω να επισέδω σε λεπτομέρειες. Το πέρασμα στο RTB Απαγορεύεται αυτό. Δεν μπορούμε να πάμε στο σύστημα legacy. Υπάρχουν 7 μόνο για το θαλής. Υπάρχουν πολλά συστήματα. Από τα πολλά εθνικά συστήματα θα περάσουμε σε ένα ευρωπαϊκό. Δεν θέλουμε το TB, το TB+, Δεν είναι αυτό το ερώτημα πώς θα περάσουμε το ένα στο άλλο. Το RTMS θέλουμε να λειτουργήσει σωστά. Και να ανταλλάξουμε εμπειρίε. Και να είμαστε σίγουροι ότι η έκδοση 3 ευθύ εξ αρχής θα εμπεριέχει όλα τα, όλες τις διορθώσεις, τα προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσει κατά το παρελθόν. Με έκπληξη διαπιστώνουμε τεράστια διαφορά όσον αφορά τη διαχείριση των συστημάτων οι χειριστές υποδομών δεν μιλάνε απαραίτητα με τις υδρομικές επιχειρήσεις. Το ξέρουμε αυτό. Τώρα τι κάνουμε. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Η ομάδα συντονισμού πρέπει να καταβάλει τις προσπάθειες για να ενταχθούν αυτά που πρέπει τα στοιχεία στο σύστημα που θέλουμε να επιβάλλουμε. Κύριε Βαντάλεν, να επιστρέψω στο θέμα της ασφάλειας όσον αφορά τους εμπορικούς σιδηροδρόμους, τι εμπορικέ αμαξοστοιχίε. Είναι το θέμα της ασφαλείας σημαντικό για μα. Στην περίπτωση του Βιαρέτζο, εκεί θεωρήσαμε ότι ήταν αποτέλεσμα τη φιλελευθερωποίηση. Δεν αληθεύει αυτό. Οφειλόταν σε ένα παλιό σύστημα που βασιζόταν στου παλιού κανόνε και έχει σε νέου κανόνε. Το νέο σύστημα, στο νέο σύστημα έπρεπε να υπάρχει σύστημα διαχείριση ασφάλεια από πλευρά της εταιρεία. Αυτά που υπόθηκαν για το Διαρέτζο τελικά απήχαν πόρο της αληθείας. Το εξετάζουμε προσεκτικά το θέμα με εμπειρογνώμονε, με τι εθνικέ αρχές. Και γίνεται συνεχή ανταλλαγή ε, πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων φορέων. Και σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές και όχι αρνητικές. Δυστυχώς, το, μεγάλο, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε στα περισσότερα κράτη-μέλη, είναι η ανάλυση των ε, ε, δυστυχημάτων. Γιατί πολλές φορές μετά από ένα δυστύχημα θεωρούνται τα συστήματα ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνα από ότι είναι. Το ERME είναι το κέντρο ερευνών. Εκεί συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, τα θέματα των αρμοδιοτήτων. Ο κύριος ε, Κράμερ το έθεσε το θέμα. Η υπηρεσία εκτελεί τις ανατεθήσει αποστολέ. Έχουμε νομικό πλαίσιο που μας επιτρέπει να εκτελούμε τις αποστολές που μας έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα. Κάτι που διαπιστώσαμε στη διάσκεψη του Διαρέτζου είναι ότι όλε οι αρχέ, οι εταίροι, θέλουν να παίρνουμε περισσότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Περνάμε μεταβατική περίοδο, νέα οδηγία, στις 19 Ιουλίου, επομένου έτους θα ισχύσει. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα. Το να αλλάζει μια νομοθεσία πριν αυτή ακόμα εφαρμοστεί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει προσπάθειες να καταβληθούν σε μεσοπρόθεσμη στόχευση. Να πούμε, το επόμενο στάδιο θα είναι αυτό. Για την ώρα έχουμε κάποια σημαντικά καθήκοντα και αγράφησα το επόμενο βήμα την ενίσχυση του ρόλου της υπηρεσίας έναντι των εθνικών ομάδων ασφαλείας αλλά με το σημερινό νομικό πλαίσιο έχουμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις ανατεθήσεις αποστολές θα έλεγα ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα να τα συζητάμε αυτά όταν κατατίθεται ο προπολογισμό για το περιβάλλον. Αυτά που πετύχαμε δεν είναι τόσο ορατά. Θα το συζητήσουμε αυτό αύριο στη Σουηδία. Σε κάθε μία από τις δραστηριότητές μας έχουμε εισάγει κάποια στοιχεία στα STI για το υλικό που χρησιμοποιείται στους υδροδρόμους, το κινούμενο, έχουμε συμπεριλάβει διάφορα στοιχεία που είναι ευνοϊκά για το περιβάλλον. Δεύτερον, το περιβάλλον δεν συνδέεται άμεσα με τις αρμοδιότητές μας, είναι κάτι που αφορά περισσότερο άλλο φορέα. Ο ίδιος ο τομέας, όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, όσον αφορά το φρενάρισμα, θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες. Να δει τι ίχνος αφήνει ο τομέα στο περιβάλλον. Δεν έχουμε οριζόντιες δραστηριότητε όσον αφορά το περιβάλλον. Συμπεριλαμβάνουμε το περιβάλλον σε διάφορα κείμενα. Προσωπικά είναι από τους τομείς στους οποίους, οποίους θα έπρεπε να αναπτυχθεί η υπηρεσία. ο άλλο φορέα που ήταν το περιβάλλον δεν είχε τα αναγκαία μέσα να υλοποιήσει περιβαλλοντικού στόχου. Όσον αφορά εν γέννη τεχνικέ πτυχέ, θα μπορούσαμε να κινηθούμε προ την κατεύθυνση του περιβάλλοντο και πιστεύω ότι αυτό θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο. Ευχαριστώ. Έχουμε κάνα δύο ερωτήσεις και έχουμε περίπου ένα 20 λεπτό. Καταλαβαίνω βέβαια ότι είναι καλές οι πληρέστατες απαντήσεις, λάβετε όμως υπόψη και το χρόνο και το σφυρί που κραδένω. Ο κύριος Πακ είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ερώτημα. Συμμερίζομαι την άποψη του Βανσκίπ όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Όμως υπάρχουν προβλήματα, κυρίως στα συνοριακά σημεία, στα σύνορα των διαφόρων χωρών. Υπάρχουν εθνικοί κανόνες περισσότερο που επικρατούν εκεί. Τι προπτική υπάρχει για μια εναρμόνιση των κανόνων αυτών. Θα μπορούσε κάτι να γίνει ή θα είναι πάντα αρμοδιότητα των Εθνικών Φορέων Ασφαλείας. Υπάρχει η δυνατότητα εναρμονίσεως. Υπάρχει η δυνατοτητα εναρμονισεως υπαρχει δυνατοτητα εκ των υστέρων ελέγχου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ουγγιάς. Eh, Δύο ερωτήσει. Στην παρέμβασή σα, αναφερθήκατε στη δραστηριότητα μελέτης και ανάλυση όσον αφορά κυρίω τα εθνικά δίκτυα και τοπικά και περιφερειακά δίκτυα. Μπορείτε να μας πείτε κάτι όσον αφορά τα κριτήρια και την όλη προβληματική που εξετάσατε και που είδατε. Δεύτερον, ερώτημα για την ασφάλεια και επιστρέφω όσον αφορά την τραγωδία της 29ης Ιουνίου την τραγωδία του Βιαρέτζο. Όσον αφορά την υπηρεσία, αυτό ήταν ε, μια σημαντική δοκιμή. Δεν ήθελα να ξέρω αν δώσατε προσοχή όσον αφορά τη διαπίστωση των επιπέδων ευθύνης. Υπάρχει κάποιο στοιχείο που εντοπίσατε μέσω δραστηριοτήτων οι χειριστές του δικτύου, οι χειριστές των σιδηροδρομικών, των αμαξοστοιχειών, οι χειριστές των εμπορευμάτων, πού εντοπίζονται οι ευθύνες. Μετά, ποια ήταν τα προβλήματα όσον αφορά τον εντοπισμό των διαφόρων αρμοδιοτήτων. Αρμοδιότητα της υπηρεσίας και αρμοδιότητα των εθνικών υπηρεσιών. Muchas Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αφού σας άκουσα, κατά πόσον γνωρίζετε το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό συνδιοδομικό Δίκτυο, ένα Ευρωπαϊκό Ανταγωνιστικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο Μεταφοράς ε, Εμπορευμάτων. Με την εισήγηση που κάνατε, με τα προβλήματα που έχουν τα δίκτυα που διαχειρίζεστε, τι, πώς κρίνεται αυτό το νέο σχέδιο. Ακούσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά δίκτυα με προβλήματα και ασφάλειας μεταξύ άλλων. Μέχρι ποιο, ποιο επίπεδο είναι συμπληρωματικά. Τα δίκτυα που περιλαμβάνονται στο παράδειγμα του σχεδίου που σας αναφέρω έχουν κάποια σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο κολλάνε και για να άποψή σα, τι προβλήματα θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτό το νέο σχέδιο οικονομισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Λιμπεράτσικη. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση έτσι λιγάκι για να τη σκεφτούμε. Κάποια στιγμή θα τελειώσει η κρίση στην Ευρώπη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς ε, πώς πιστεύετε ότι θα βγούμε από αυτή την κρίση ως ε, σιδηρόδρομοι. Δηλαδή έχουμε άραγε κάποια δυνατότητα να καταλάβουμε μια νέα θέση ε, σχετικά με το που θέλουμε να προχωρήσουν οι σιδηρόδρομοι ή θα παραμείνουν όλα παράλλαχτα. Αν δεν υπάρχει κανείς άλλος θα μου επιτρέψετε να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Ο εισηγητής ε, εξέφρασε τις ανησυχίες ε, αρκετών ε, κρατών μελών σχετικά με τα εμπορεύματα στην Ευρώπη κυρίως και φαίνεται ότι είναι μεγάλο πρόβλημα το να περνάνε τα εμπορευματικά, η εμπορευματική σειρμή μέσα από ε, κάποιες χώρες χωρίς να αναπτύσσουν ταχύτητα. Ο κύριος Μπακ ε, σας ρώτησε τι θα γίνει με την εναρμόνιση. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι οι διαφορετικοί μηχανισμοί κοστολόγησης. Ας πούμε, πάρουμε από το Λονδίνο στο, στη Λίλ... Ε, πρέπει εκεί να έχει κανείς κατά νου. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές τιμές ε, ναύλη για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα των εμπορευμάτων μας ανησυχεί. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και επίσης υπάρχει και διαφορά ανάμεσα στη Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη όσον αφορά την προσφορά υποδομής, ε, και ο ορισμός του τρένου υψηλής ταχύτητας στο ανατολικό κομμάτι της Ευρώπης διαφέρει ριζικά από το τι είναι τρένο υψηλής ταχύτητας στη Δυτική Ευρώπη. Κατόπιν, ε, όσον αφορά τα εργαστήρια και το θέμα της ε, κληρονομιάς, κατά πόσον δηλαδή ε, τα εργαστήρια τα οποία ασχολούνται με αυτές τις παραδοσιακές γραμμές και κάποια στιγμή περνάνε σε μεγάλες ε, αποστάσεις. Αυτά τα μικρά τρένα καλύπτονται από την ε, οδηγία για ασφάλεια. Δηλαδή, ξέρω πολύ καλά ότι εξαιρούνται αυτές οι ειδικέ γραμμές ε, που έχουν σχέση με την προστασία της κληρονομιάς, αλλά εν πάση θέλω να γνωρίζω τι ακριβώ συμβαίνει σε περιπτώσεις ε, μεγαλύτερων τρένων. Κυρίως όταν χρησιμοποιείται τροχαίο υλικό σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, υπάρχει ένας κατάλογος ε, όλων των εθνικών μέτρων ασφαλείας ε, και τεχνικοί κανόνες. Είναι η νέα δραστηριότητα του cross acceptance που θα παρουσιαστεί και αύριο στα πλαίσια ενό εγγράφου αναφορά αποτελεί το πλαίσιο του όλου ενίγματο. Διότι όλοι οι κανόνε αποτελούν ένα ένιγμα, ένα μοσαϊκό. Υπάρχουν οι κανόνε ασφαλεία, οι τεχνικοί κανόνε, οι άγνωστοι κανόνε που αποκαλούνται, οι μη, οι μη εφαρμόσιμοι κανόνε κλπ. Αυτοί που δεν εφαρμόζονται μάλλον. Λοιπόν, υπάρχει φοβερή σύγχυση βάζει κανόνε. Στόχο είναι ένα κατάλογο κανόνων που κοινοποιούνται και να εντοπίζονται αυτοί οι κανόνε. Έλεγα στη ότι πριν μερικού μήνε και με 2 με 3-3% κανόνων που κοινοποιούνται. Σήμερα, χωρί να κοιτάμε το περιεχόμενο, είμαστε στο 50%. Προχωράει η διαδικασία. Αφού γίνει αυτό ο κατάλογο, η πραγματική προστιθέμενη αξία θα ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε σύγκριση, να δούμε ισοδυναμίε και να αποφύγουμε έτσι τα προβλήματα που έχουμε. Να υπάρχει, παραδείγματο χάρη, σε ένα τρένο υψηλή ταχύτητα, ένα πυροσβεστήρα που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη χώρα ή τα πρώτων βοηθειών που διαφέρουν, τα κουτιά πρώτων βοηθειών που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αυτό είναι το έργο τη πολλαπλή αποδοχή του cross acceptance, συσσόρευση, συγκέντρωσης, σύγκριση. προχωράμε πολύ γρήγορα και θέλουμε να μα δοθεί εντολή αρκετά ευρεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσον αφορά το θέμα. Τι διαπιστώνουμε πολύ συχνά είναι ότι οι κανόνε είναι ταυτόσιμοι, οι αρχέ, είναι ισοδύνας χρησιμοποιούνται, αλλά όλοι θα έπρεπε σε κάθε διέλευση συνόρων να κάνει την επαλήθευση όταν αυτό δεν χρειάζεται. Εκεί θα ήταν η προστιθέμενη αξία τη ε, ε, δουλειά μα, να πρέπει να έλεγχοι. Όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με τα δίκτυα, σήμερα οι κανόνε μα εφαρμόζονται σε όλο το διευρωπαϊκό δίκτυο, σε όλο το τροχαίο υλικό βέβαια και ε, στο αυτούς που είναι εκτός διευρωπαϊκών δικτύων, δηλαδή Πρέπει να εφαρμόζονται τα STI, χρειάζονται όμω οι εταίροι και τα κράτη-μέλη να καθορίσουν ποια τα δίκτυα καλύπτονται από του κανόνε του εφαρμοστικού και ποια δίκτυα, δίκτυα εν μέρη και ποια δίκτυα απαλλάσσονται ή εξαιρούνται. Όπω ιστορικέ ε, συνδρομικέ διαδρομέ. Όπω αφορά το ατύχημα του Βιαρέτζο, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Σήμερα δεν έχουμε την έκθεση της Εθνικής Αρχής Έρευνας. Φυσικό είναι αυτό. Δεν έχουμε λοιπόν αυτή την έκθεση από την Ιταλία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να λάβουμε αυτή την έκθεση ε, του οργανισμού έρευνας από τι φοροτιμής στη δουλειά της εθνικής, την Ιταλική υπηρεσία, Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας που συνεργάζεται στενά με μας ε, δίνει στοιχεία, παραδείγματο χάρη το είδος των αξώνων, τέλος πάντων διάφορα τεχνικά στοιχεία σε άλλους συνδρομικού φορεί άλλων χωρών για να μπορούν να γίνουν εξακριβώ επαληθέ συγκρίσει. Ποτέ δεν έχει μία αιτία ένα τύχημα. το χάρη μπορεί να έχει σπάσει ένα άξονα, μπορεί να έχει χαλάσει κάποιο ανταλλακτικό, κάποιο στοιχείο. Διάφορα παίζουν ρόλο σε ένα τύχημα. Δεν από πλευρά του Ιταλικού φορέα. Και αυτό σημαντικό παρόλο που μας ζήτησαν υποστήριξη. Και παρακολουθούμε καθημερινά τις προσπάθειες. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα όταν δεν έχουμε τα συμπεράσματα του οργανισμού έρευνες, όπως είπα πολλές φορές. Το θέμα είναι κατά πώς υπάρχει πρόβλημα αρμοδιοτήτων μεταξύ της υπηρεσίας και των εθνικών αρχών. Λοιπόν, για την ώρα όχι. Αντίθετα, οι σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές, διότι όλοι είμαστε παιδιά του δεύτερου πακέτου και πάνω απ' όλα έχουμε αναπτύξει όλοι νέα συστήματα. Βγαίνουμε από ένα αυτορυθμιζόμενο σύστημα προς ένα σύστημα πάμε που ρυθμίζεται από άλλους ε, φορείς και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Καμιά φορά η απελευθέρωση του τομέα των σιδηροδρόμων μπορεί να γίνει απελευθέρωση, άνοιγμα, αλλά είναι πολύ δύσκολη αυτή η μετάβαση. Είναι καλές οι σχέσεις, ίσως Καμιά φορά θα ενισχυθούν οι, ρόλοι. Θα το συζητήσουμε αυτό. Τι είναι το θετικό. Όλες οι εθνικές αρχές ασφάλειας δέχτηκαν την πρόταση που έκανα την επομένη της διάσκεψης του Βιαρέτζου, δηλαδή ε, να υπάρξει μια δομή προβληματισμού που θα ενισχύσει ίσως και το δικό μας ρόλο και το δικό τους ρόλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί με τον ίδιο ενθουσιασμό ευρωπαϊκά δίκτυα. Το νέο δίκτυο έχει το πλεονέκτημα ότι είναι νέο ακριβώ, κύριε μου, και πρέπει να πληρεί τι νέε τεχνικέ προδιαγραφέ που έχουμε θέσει. Άρα, εξ ορισμού θα ε, διαμορφωθεί με βάση του όσο περισσότερο μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα γίνεται. Αυτό είναι ήδη θετικό. Επίσης να σα πω ότι στον τομέα αυτό όπω και αλλού πρέπει να φροντίσουμε ούτω ώστε οι επενδύσει που γίνονται να τηρούνται με να τηρούν τις προδιαγραφές αυτές. Κάτι δεν συμβαίνει πάντα. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθήσουμε και τις εργασίες στους μεγάλους διαδρόμους, στα μεγάλα έργα. Γιατί βλέπουμε ότι μερικοί ευρωπαϊκοί κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται δεν πολύ εφαρμόζονται ανά Είναι φανές ότι το δίκτυο Μάλλον ένα από τα προβλήματα ανάπτυξης των εμπορικών μεταφορών είναι η, το, η χωρητικότητα. Ε, ε, το παράδειγμα του Βελγίου είναι κλασικό παράδειγμα επιπλέον έχουμε, δεν έχουμε αρκετά, ε, αρκετές αμαξοστοιχίες μετακίνηση ε, για τις μανούβες, κάτι που είναι βασικό πρόβλημα. Σε ό,τι μας αφορά δεν μπορούμε να λάβουμε θέση και να γνωμοδοτήσουμε σε σχέση με μια συγκεκριμένη γραμμή ή ένα συγκεκριμένο δομολόγιο. Η άποψή μας είναι ε, αυτό μπορεί να πούμε είναι τηρεί του τεχνικούς κανόνε ή όχι, είναι διαλειτουργικό ή όχι, πληρεί τους κανόνες ασφαλείας, αλλά όχι να κρίνουμε αν είναι ε, σωστή ή όχι μια γραμμή, αν πρέπει να συνεχιστεί ή όχι. Αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Εμεί έχουμε μια ε, δυνατότητα να πούμε και αυτό το λέει και το ευρωπαϊκό το σχέδιο μνημονίου συνεννόηση που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ότι ναι, τηρούνται οι κανόνε διαλειτουργικότητα, οι κανόνε ασφάλεια. Δύο ακόμα. Το charging. Δεν έχουμε ευθύνη για το charging, πρόεδρε, για την τιμολογική πολιτική. Είναι θεωρήσει. Διαφορέ μεταξύ Ανατολική και Δυτική Ευρώπη σε όλου του υπάρχουν ε, στην Ανατολική Ευρώπη υπάρχουν πολλές ε, ευθύνες, πολλές θερμοδιότητες. Δεν είμαστε ωστόσο τυφλοί. Είχαμε μια συνάντηση πριν από λίγες μέρες με τον κύριο Μαζάτσα στα, στα κρατημέλη και ήταν προφανές ότι η οικονομική κατάσταση των οργανισμών είχαν συνέπειες στην ασφάλεια. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι προσπαθούμε να ορίσουμε την κοινή θέση με βάση τους κανόνες, αλλά είναι σαφές ότι είναι ένα πρόβλημα. Τι θα γίνει όταν ο σιδομικός τομέας ε, ξαναπάει τα πάνω του, καταρχάς ε, συνολικά βρίσκεται σε φάση ανάπτυξη ακόμα, όχι για τις εμπορευματικές μεταφορές, ε, συνολικά. Επιβατικές, το χείο Τώρα ένα υψηλή ταχύτητα αναπτύσσονται ακόμα και χρειάζεται και ανανέωση του υλικού, αλλά είναι σε ανάπτυξη. Δεύτερο θέμα που θέλω να τονίσω. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι όλα να γίνονται με βάση τυποποιημένα συστήματα. Να υπάρχει δηλαδή εμπιστοσύνη λέγοντα ότι εγώ επενδύω στο ETMS e γιατί είναι σωστό και αξιόπιστο σύστημα, ότι θα υπάρχει γρήγορη και φθηνή πιστοποίηση. Αυτό είναι σημαντικό για τις εθνικές αρχές. Και η πρόκλησή μας είναι αυτή. Έχουμε δύο-τρία χρόνια μπροστά μας σήμερα για να ολοκληρώσουμε. Για όταν λέω ολοκληρώσουμε εννοώ εμείς και ο κλάδος. Το παζλ που σας έδειξε προηγουμένως.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 Κυρίες και κύριοι, είμαι ο επικεφαλής ε, της ε, ομάδας ασφαλείας, ε, της μονάδας ασφαλείας για τους ευρωπαϊκούς σιδηρόδρομους και αναφέρομαι κυρίως στα εργαστήρια συντήρησης και για τα ιστορικά δρομολόγια και για τα κανονικά. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο φορέας μας σχετικά με αυτά τα εργαστήρια συντήρησης δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα, δουλεύουμε, προετοιμαζόμαστε και θα είμαστε έτοιμοι μετά από κάποιους μήνες. Τώρα, όσον αφορά την προσέγγιση, η προσέγγιση μας ε, είναι προαιρετική. Εναπόκειται λοιπόν στο ίδιο το εργαστήριο να ζητήσει πιστοποίηση ή όχι. Πάντως, καταρτίζουμε επίσης και ένα σύστημα πιστοποίησης για φορείς που είναι αρμόδιοι για τη συντήρηση, όπως αναφέρεται και στην ορολογία της νέας οδηγίας. Δηλαδή ένας φορέας που θα αναλαμβάνει πλήρως ε, τη συντήρηση, μακροπρόθεσμη συντήρηση ενός ε, σειρμού και αυτό λοιπόν το σύστημα θα είναι δεσμευτικό με βάση την ε, τροπολογία που κατατέθηκε για την οδηγία ασφάλειας. Βεβαίως το εργαστήριο ε, μπορεί να παραμείνει, αυτό δεν το αποκλείουμε και στην περίπτωση αυτή η πιστοποίηση θα είναι δεσμευτική και για ένα εργαστήριο που θα συνδυάζει τους ιστορικούς σιδηρόδρομους ε, και τους κανονικούς ε, βαριούς σύρμους. Εξαιρούνται βέβαια κάποιοι σειρμοί από την εφαρμογή της οδηγίας. Ελπίζω να ήμουν σαφής και να απάντησα στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε, ε, ξέρω βέβαια, είναι δική μου οδηγία σχετικά με την εξαίρεση. Υπήρχε κάποια επικάλυψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που ήρθατε για να μας απευθύνετε το λόγο. Όλα αυτά αποτελούν κομμάτι αυτών που ασχολούμεθα με τους ε, διάφορους φορείς ε, για τους σιδηρόδρομους. Ασχοληθούμε, ασχοληθήκαμε με την αεροπλοία, θα ασχοληθούμε αύριο και με την αυτιλία, έτσι ώστε όλα τα μέλη, κυρίως τα νέα μέλη, να ενημερωθούν για τους ε, φορείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και προσβλέπουμε στο να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία μαζί σας. Thank you. Thanks a lot. So, next item is the European... Λοιπόν, επόμενο θέμα είναι το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές. Είστε έτοιμος κύριε Μαρινέσκου. Μάλιστα. Πανέτοιμος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, ψήφισε το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο σε πρώτη ανάγνωση για αυτό τον κανονισμό. Ε, το Συμβούλιο ψήφισε τον Ιούνιο και εκεί συμφωνήσαμε επί του κειμένου. Εγώ λοιπόν υιοθέτησα την έκθεση αυτή στη συνεδρίαση ε, υιοθέτησα την έκθεση αυτή τον Αύγουστο και συναντήθηκα με εκπροσώπους ε, της Επιτροπής ε, και του Συμβουλίου. Και μπορώ να σας πω ποια θα είναι τα βασικότερα θέματα που θα συζητηθούν όσον αφορά αυτόν τον κανονισμό. Πρώτον, επιγή των διαδρόμων η διάσταση απόψεων στα τρία διαφορετικά κείμενα στο αρχικό κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εκεί υπάρχει μια ε, εναλλακτική λύση όπου τα κράτη-μέλη μετά την έγκριση του κανονισμού καλούνται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αποφασίσουν τουλάχιστον για ένα διάδρομο που θα διασχίζει ένα κράτος μέλος. Άλλοι πάλι λένε ευθύς εξ αρχής να καθοριστεί συγκεκριμένος αριθμός ε, διαδρόμων και αυτό με τη μορφή παραρτήματος στο συγκεκριμένο κανονισμό. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε Αυτά που προτείνει το Συμβούλιο καλύπτουν τόσο την πρόταση της Επιτροπής όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε ότι αν τελικά υπάρχει, υπάρξει παράρτημα θα συμπεριληφθούν όλα τα κράτη-μέλη και κυρίως εκείνα τα οποία διαθέτουν σιδηροδομικό δίκτυο. Κατόπιν, επίμαχο θέμα, επόμενο επίμαχο θέμα. Αυτός ο διάδρομος τι είδου διαχείριση ε, θα την χάνει. Ναι, μεν προβλέπεται κάποιο φορέα διαχείριση ε, και κάποιο ευρωπαϊκό οργανισμό. Τώρα το Συμβούλιο προτείνει να συστηθούν δύο φορείς, ε, ένας διαχείρισης και ένας τεχνικός που θα αποτελούνται από τις ε, ανάλογες ε, δομές διαχείρισης ενός κράτους ε, μέλους που ασχολούνται με τους διαδρόμους. Νομίζω και εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε, μπορούμε να επιτύχουμε συμβιβασμό. Το τρίτο θέμα αφορά την προτίμηση. Η πρόταση Κομισιόν εκφράζει την προτίμησή της για τις εμπορευματικές μεταφορές. Το Κοινοβούλιο είπε ότι σε περίοδους εχμής προτεραιότητα πρέπει να έχουν ε, η ε, επιβατική σειρμή επιβατών. Νομίζω, μπορούμε βέβαια να ισχυριστούμε ότι προτεραιότητα μπορούν να έχουν και τα εμπορεύματα, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Και τέλος, ε, One Stop Shop, εκεί νομίζω οι διαφορές είναι πολύ περιορισμένες δεν θα υπάρξουν πρόβληματα και ε, θα επιτύχουμε ταχύτατα συντονισμό. Η κατάσταση λοιπόν είναι η εξής. Το το Συμβούλιο ε, μπορεί να μας ε, διαβιβάσει την πρόταση του αρχές Δεκεμβρίου. Η Σουηδική Προεδρία επιθυμεί να ολοκληρωθεί το θέμα εφέτος. Ενδέχεται λοιπόν στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου να επεξεργαστούμε το συγκεκριμένο κείμενο. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάρουμε την εντολή για να επιτευχθεί η συμφωνία μέχρι το Δεκέμβρη, έτσι ώστε το Δεκέμβρη το Συμβουλίο να μπορεί να κρίνει ένα κείμενο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να θεσπίσει Ιανουάριο-Φεβρουάριο ε, το κείμενο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή δυνατότητα για να προχωρήσουμε. Τα τόπιν. Όσον αφορά τώρα ε, τους ε, οι εισηγητές ε, και τους και συγητές όλα έχουν ε, οριστεί και μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Σουηδική Προεδρία για να ολοκληρώσουμε το θέμα το Δεκέμβρη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λιμπεράτσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέσκου συνεργαστήκαμε στενά μαζί. Ε, συναντήσαμε εκπροσώπους του Συμβουλίου και τους κοιοδησηγητές. Είμαστε αρκετά ανοιχτοί στις θέσεις για τις διαπραγματεύσεις. Γιατί μερικέ φορέ ε, τίθενται και ορισμένα θεωρητικά ερωτήματα. Γιατί χρειαζόμαστε τον κανονισμό αυτό, τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτόν, ιδίω όταν ε, λέμε ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα των συνδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη. Για κάποια χρόνια είχαμε την οδηγία απελευθέρωση των συνδρομικών μεταφορών, δεν έγινε ωστόσο τίποτα το σημαντικό στον τομέα αυτό. Υπάρχει ένα δίλημα. Θα έπρεπε να αγωνιστούμε για τους διαδρόμους αυτού με τις χώρες να δώσουν τους διαδρόμους, γιατί μερικές φορές δεν θέλουν να δηλώσουν ότι είναι έτοιμοι να παράσχουν ένα τέτοιο διάδρομο. Γιατί? Γιατί συχνά απαιτεί επενδύσεις, δουλειά, οικονομική και ε, υποδομή. Η άποψή μου λοιπόν είναι εξή. Οι χώρε που ενδιαφέρονται θα έπρεπε να μπορούν να το κάνουν. Προφανώ βέβαια δεν χρειαζόμαστε πολλού διαδρόμου. Καλύτερα να έχουμε λίγου και καλού που να λειτουργούν εκεί που μπορεί να λειτουργήσουν και να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν εκεί που είναι δυνατό. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Επιτροπής. τους φορείς διαχείρισης. Τι θα διαχειρίζεται αυτός ο φορέας διαχείρισης. Αφού δεν θα μπορεί να αποφασίζει για την τιμολογιακή πολιτική, τον άβλο θα τον καθορίζει το εθνικό όργανο. Αυτή η μονάδα διαχείρισης δεν θα δίνει σλότ σιδηροδρομικά, ας πούμε, ούτε θα αποφασίζει για το ποιος θα έχει αυτά τα σλότ και αυτά θα αποφασίζονται από τις εθνικές αρχές που διαχειρίζονται το, κάθε σύστημα. Αυτή η μονάδα λοιπόν διαχείρισης, τουλάχιστον έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν θεωρούμε ότι είναι μια μονάδα που εναρμονίζει το οτιδήποτε πρότυπα ε, σε ό,τι αφορά την ομογενοποίηση της ε, των άβλων των της τηλεμοριακής πολιτικής. Ούτε θα επιβάλλει πρόστιμα, ας πούμε, σε εταιρείε που έχουν δεσπόζουσα θέση. δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός. Άρα το κατασκεύασμα αυτό δεν... Το, μάλλον το κατασκεύασμα αυτό σήμερα δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο στην ομάδα διαχείρισης. Υπάρχουν βέβαια μονάδες όπου συναντούνται οι και όπου θα, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα βήμα μπρος. Και θα δίνουν σλότς. Στο μέλλον όμως, όχι τώρα, όπως για τις αερομεταφορές. Θέλουμε να αναζητήσουμε, να δημιουργήσουμε μια αντίστοιχη κατάσταση. Αλλά πραγματικά το χρειαζόμαστε. Χρειάζεται να διαμορφώσουμε κάτι τέτοιο ή μήπως αρκεί να αφήσουμε τις αγορές να ρυθμιστούν μόνες τους. Και δεν χρειάζεται να υπάρχουν ε, δηλαδή να περιμένουμε τρία-τέσσερα δίκτυα να, να, αποφασίζουν για την τελική τιμή. Στη δική μου πολιτική ομάδα πιστεύουμε ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στα επιβατικά τρένα. Γιατί μιλάμε εκεί για ανθρώπους. Και όταν μιλάμε για επιβατικές μεταφορές μπορεί να παράσεις ένα χρονοδιάγραμμα μήνες πριν. Αν περιμένει ένα εμπορικό τρένο δύο ώρες, δεν είναι πρόβλημα. Αν περιμένει ένα τρένο με επιβάτες δύο ώρες, είναι. Ελπίζω ότι θα παρέχουμε Ελπίζω να δώσουμε μια σωστή εντολή για να, στον ε, εισηγητή μας για να προχωρήσει. Κύριε Μπιλμπάο, ευχαριστώ. Μεταξύ των σημείων που υπογράμμισα που υπογράμμισε ο κύριος Μαρινέσκου θα επαναφέρω κάτι που είπα και σε άλλες συναντήσεις που είχαμε. Μιλούμε για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο και αντί να συζητούμε ποιο διάδρομο θα, σε ποιο δρόμο θα δώσουμε προτεραιότητα και σε ποιον όχι. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε σαφή εικόνα των κριτηρίων, των σαφών κριτηρίων που οδήγησαν το Συμβούλιο να ορίσει στο παράτημα τα οκτώ, τους εκτό νέους διαδρόμους. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποια γραμμή θα σχεδιάσουμε, τι επιπτώσεις θα έχει ο σχεδιασμός αυτός στα υπόλοιπα δίκτυα που είναι στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να ξέρουμε με τα έργα αυτά ποια σημεία σύγκρουσης ή κορεσμού θα λύσουμε με τους νέους διαδρόμους. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για το πώς διαχειριζόμαστε ένα διάδρομο, ποιες προτεραιότητες δίνουμε, ποιες πιέσεις υπάρχουν και πώς θα καταλήξουμε στην, ε, στο, ε, εν, στο ενιαίο στην ενιαία λειτουργία. Πρώτα όμως πρέπει να δώσουμε τον ορισμό του ευρωπαϊκού σχεδίου. Τι στόχο έχουμε, τι σαφή στόχο έχουμε με τα, τους διαδρόμους, τι θέλουμε να πετύχουμε τώρα, τι θέλουμε να λύσουμε και τι εγχείρημα θα κάνουμε, ούτως ώστε αυτό να είναι καλό για όλους τους Ευρωπαίους. Με μια σελίδα αρκούσε κάτι τέτοιο. Ένα σχέδιο, τι υπάρχει, τι προβλέπεται και τι λύνουν οι νέοι διάδρομοι. Αυτό θα ήταν χρήσιμο για να μπορέσουμε εμείς στην Επιτροπή τουλάχιστον να έχουμε μια εικόνα της νέας κατάστασης. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριος Κρέμερ.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 Κοιτάξτε, ε, υπάρχει έκφραση ε, συνονθήλευμα εθνικών εγωισμών. Ε, αυτό όμως δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με την πολιτική μεταφορών. Κοιτάξτε, έχουμε ήδη έξι διαδρόμους για το ERTMS, κυρίως για τις εμπορευματικές μεταφορές. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους έξι διαδρόμους. Αυτοί υπάρχουν πάνω από δέκα χρόνια και από αυτούς κανένας όμως ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Πιστεύετε ότι τώρα αν ανοίξουμε και άλλο διαδρόμο όμως τα πράγματα ε, θα προχωρήσουν γρηγορότερα, κάθε άλλο. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτός ο ERTMS ε, ακόμα δεν είναι έτοιμος. Ε, στη Γερμανία κανείς δεν έχει πάρει ακόμα το κομμάτι του Ρήνου, παρότι ξέρουμε ότι αυτό το κομμάτι είναι το πιο σημαντικό στην Ευρώπη. Και τι κάνουμε τώρα, ασχολούμαστε με νέους διαδρόμους. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, ποια είναι τα κίνητρα τα κίνητρα είναι η εθνική περηφάνεια των κρατών μελών αν είναι εγωιστές, τότε πρέπει και να του ρωτήσουμε και μέχρι ποιο σημείο θα χρηματοδοτήσετε. Αν είχαμε ορίσει συγκεκριμένα ποσά χρηματοδότησης, τότε θα μπορούσα να το δεχτώ και να πω εντάξει, αν ο πέμπτος ή έκτος σιδηρόδρομος δεν προχωράει, ας έρθουν άλλοι, ας προχωρήσουν άλλοι. Τώρα όμως ε, το να προσθέσουμε άλλους 5-6 που καθυστερούν, αυτό δεν αλλάζει τίποτα στους ε, ευρωπαϊκούς ε, όρους και προοπτικές. Ως εκ τούτου, εγώ θεωρώ ότι πρέπει τώρα να επεκταθούμε, δεν, δεν πιστεύω ότι θέλουν να επεκταθούμε σε, στους 9. Παραδείγματος χάρη, ο υπαριθμόν 3. Αυτός αναφέρεται από, το Στοκχόλμο, από τη Στοκχόλμη στο Παλέρμο. Μάλμε, Κοπενχάγη, Αμβούργο, μετά Μεγάλο Κενό, μετά Ινσπρουκ, Βερόνα, Παλέρμο. Ε, εν τω μεταξύ όμως ενδιάμεσα τι θα γίνει. Γιατί αναφέρεται το Αμβούργο. Παρότι η συντομότερη σύνδεση είναι Βερολίνο, Παλέρμο και η ε, πιο σύντομη ε, διαδρομή είναι μέσα από τη, από τη Ρόστοκ. Ε, και ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αν ε, θα υπάρξει σύραγγα ή ε, γέφυρα, αν θα μπορεί να περάσει ο σιδηρόδρομος από εκεί, όχι. Κοιτάξτε, πρέπει να ξέρετε το εξή. Εδώ βάζουμε προτεραιότητε που θα υλοποιηθούν μετά από 20 χρόνια. Δεν υπάρχει καμία επιτάχυνση. Και γιατί δεν γίνονται όλα αυτά. Παράλληλα, αν πάρουμε τις χώρες, Έκανα κάποιον υπολογισμό. 27 είμαστε τα κράτη-μέλη. Δύο κράτη δεν έχουν καθόλου σιδηρόδρομο, αλλά 25. Και εσείς αναφέρατε 22, όχι 3. Φινλανδία, Εστονία και Λετονία. Από την άλλη έχουμε την Rail Baltica που πάει από τη Βαρσοβία στο Ελσίνκι. Και εκεί συμπεριλαμβάνονται αυτές οι τρεις χώρες. Λοιπόν, ε, στο Project αυτά δεν παίζει κανένα ρόλο η προτεραιότητα. Δηλαδή οι χώρε είπαν ε, ότι οι εμπορευματικέ μα διαφορέ μας είναι παντελώ αδιάφορε, παρότι οι γραμμέ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και από επιβατηγά τρένα και από εμπορευματικά. Γιατί δεν συμμετέχουν αυτές οι τρεις χώρε σε εμπορευματικές μεταφορές ενώ στο πρόγραμμα των προτεραιοτήτων αναφέρονται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό ε, πρέπει να εξηγηθεί ίσως ε, και να ήταν ιδιαίτερη τίμη και να λένε λόγω της οικονομικής κρίσης έχουμε τεράστια οικονομικά προβλήματα. Τότε όμως και εγώ διερωτώ με οι άλλες χώρες δεν θίγονται από την κρίση και λένε «Α, ωραία, εμείς θα χρηματοδοτήσουμε σιδηρόδρομους και διαδρόμους». Αυτό πρέπει εδώ να το ορίσουμε. Για το Συμβούλιο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό όραμα, είναι απλά εθνική ανοησία. Μετά, αναφερθήκατε στο φορέα, body. Χρειαζόμαστε μια ενιαία θηρίδα για το διάδρομο υπαριθμών 1. Αν θέλει κάποιος να πάρει ένα σλότ, ε, τρεις χώρες λένε ναι και η τέταρτη λέει όχι, δεν γίνεται για εθνικούς λόγους. Πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό φορέα, ο οποίος ε, σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς ε, θα αποφασίζει για τα σλότ. Τώρα, όσον αφορά τις προτεραιότητε, εγώ είμαι υπέρ τη ευελιξία. βεβαίω και δεν πρέπει να ή υποτιμούνται οι μεταφορές ατόμων. Αλλά ε, αν υπάρξει κάποιο ατύχημα, αυτό που παίζει ρόλο είναι το συντομότερο δυνατόν να επανέλθει η κανονική κυκλοφορία. Παράδειγμα, έχουμε έναν ε, μηχανοδηγό ε, στις εμπορευματικές μεταφορές που έχει ένα τέταρτο διάλειμμα. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί αν υπάρξει τώρα ένα τρένο που έχει ατύχημα, ε, θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Όχι να κάνει διάλειμμα, να το ξεχάσει το διάλειμμα. Άρα δηλαδή ε, χρειαζόμαστε ευελιξία. Γιατί αν δεν υπάρχει ευελιξία θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Κατά τα άλλα, η άποψή μας είναι ότι χρειαζόμαστε αυτό, αυτή την ενιαία θηρίδα γιατί εμείς ε, συγκρινόμεθα ως Ευρωπαίοι. Και πολλοί λένε ότι ε, τα τρένα είναι το τελευταίο εθνικό στοιχείο που υπάρχει στην Ευρώπη. Βλέπω πολύ συμφωνείτε. Ε, ε, πόσο, πώς μπορώ να φανταστώ ότι είστε Ευρωπαίοι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά θα ήθελα να με στηρίξετε. Ο κύριος Ζέλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση. Το Συμβούλιο, προφανώς, προσέφερε κάτι άλλο πέρα από τους εννιά διαδρόμους που γνωρίζουμε στο πρώτο παράρτημα. Στο δεύτερο παράρτημα προβλέπεται μία δίωδος για εμπορεύματα για κάθε κράτος μέλος. Και μετά ο υπουργό Μεταφορών της Λετωνίας δεν θέλει να συμφωνήσει όσον αφορά αυτό το διάδρομο για τα εμπορεύματα. Δεν συμφωνώ με τον Υπουργό Μεταφορών. Η επέκταση του 8 διαδρόμου που συνεχίζει την κατεύθυνση των βατικών σιδηροδρόμων από Ρήγα προς Κάουνας και μετά μέχρι Ελσίνκη. Χρειάζεται σωστή στρατηγική να επεκταθεί αυτός ο διάδρομος. Αν σταματήσει στη Λετωνία ο διάδρομος, τότε το εμπόρευμα μετά θα πρέπει να μεταφερθεί με φορτηγά, οδικά, για να πάει σε άλλες χώρες. Προτείνω αυτό να το δούμε από ευρωπαϊκή σκοπιά. Η Λετωνία και η Εστονία θα συμμετάσχουν δύσκολα στην ανάπτυξη αυτού του διαδρόμου, το γνωρίζω. Αλλά από μια ευρωπαϊκή σκοπιά αυτό θα έπρεπε να είναι κάτι που προβλέπεται. Ταυτόχρονα καταλαβαίνω γιατί οι λετωνικές αρχές και ο ίδιος ο Υπουργός το ίδιο συμβαίνει και Εστονία και Λετωνία προτιμούν άλλη προσέγγιση. Δηλαδή ότι οι βαλτικές χώρες μπορούν να επιλέξουν το διάδρομο που θα χρησιμοποιήσουν. Το πρόβλημα με τις βαλτικές χώρες είναι η απόσταση μεταξύ των σιδηροτροχιών, το εύρος των σιδηροτροχιών. Και μέχρι τώρα στις βαλτικές χώρες χρησιμοποιούμε το ρωσικό πρότυπο. Λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές πτυχές και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να επεκταθεί ο διάδρομος αυτός. Διαφορετικά θα υπάρξουν προβλήματα. Και θα πληγούν και τα ευρωπαϊκά διευρωπαϊκά δίκτυα. Ευχαριστώ. Η κυρία Αλβάρες. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μαρινέσκου για την έκθεσή του. Είναι σημαντική ε, και βασικό στοιχείο στο μελλοντικό ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών. Είναι δε σημαντικό σαν αφετηρία για μια ανανέωση των εμπορευματικών σειρονομικών μεταφορών στην Ευρώπη, που είναι ένα εκκρεμές ζήτημα. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε ποιότητα των επιβατηγών μεταφορών και ταχύτητα στις εμπορευματικές. Πολλές λύσεις μπορούμε να σκεφτούμε. Βελτίωση των υποδομών, γραμμή ε, των, γραμμ, των παραδοσιακών γραμμών που απελευθερώνονται γιατί χρησιμοποιείται πλέον το δίκτυο υψηλή ταχύτητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παλιά γραμμή για εμπορευματικέ μεταφορές και να διευκολυνθεί η ε, διαλειτουργικότητα με τα λιμάνια. Ε, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών με σιδηρόδρομο στην Ευρώπη και που πρέπει να σχετίζεται και με την διαχείριση ωστόσο των μεταφορών που προφανώς απαιτεί μια ενιαία απόφαση. Ε, καλά κάνετε λοιπόν κύριε Μαρινέσκου και παρουσιάζετε την έκθεση αυτή ζητώντας να υπάρχει μια συμφωνία γρήγορη γιατί πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα με εμπορευματικών μεταφορών με μες στην Ευρώπη σαν ένα κομμάτι του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφορών συνολικά. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, κ. Καστελαλότη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Um, uh, βασικά θέματα ήδη υπογραμμίστηκαν από τον κύριο Μαρινέσκου. Αυτά τα βασικά θέματα είναι η επιλογή των διαδρόμων, το θέμα της διακυβέρνησης αυτών και προτεραιότητες για τα εμπορεύματα. Ξέρετε θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την επιλογή των διαδρόμων, η θέση μας ήταν η εξής, ότι αυτή η επιλογή θα πρέπει λαμβάνει η χώρα επί τη βάση αναλύσεως της αγοράς. Θα πρέπει η επιλογή να είναι ανοιχτή και επιλογή να δικαιολογείται βάσει των αναγκών της αγοράς. Η υποβληθήσα πρόταση του Συμβουλίου δίνει μια πρώτη επιλογή διαδρόμων, ένα πρώτο κατάλογο διαδρόμων και τη δυνατότητα να προσθεθούν νέοι διάδρομοι ή να τροποποιηθούν αυτοί είναι πολιτική επιλογή. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η επιλογή δεν είναι βέλτιστη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτοί οι διάδρομοι ήδη είναι πραγματικότητα, ήδη υπάρχουν, δεν του έχουμε εφεύρει. Σε πολλές περιπτώσεις συμπεριλαμβάνουμε τους έξι διαδρόμους ERTMS, τους βασικούς άξονες μεταφοράς των εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμων. Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη και κάποιο στοιχείο όσον αφορά την επιλογή των διαδρόμων. Στόχος της προτάσεως ήταν η επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων βραχυπρόθεσμα μέσω της εισαγωγής λειτουργικών μέτρων. Το δίκτυο για τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμων δεν χρειάζεται πολλές επενδύσεις. Μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας των χειριστών των υποδομών. Γι' αυτό πρέπει να τα δούμε διαφορετικά αυτά τα δίκτυα εν συγκρίση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τα προγράμματα προτεραιότητας, όπου χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις για την επίτευξη αποτελεσμάτων μακροπρόθεσμα. Θέλουμε να πετύχουμε αποτελέσματα μέσω βραχυπρόθεσμα, διότι μόνο εντός αυτού του χρονικού περιθωρίου θέλουμε να αναζωογονήσουμε τη μεταφορά εμπορευμάτων. Όσον αφορά την διαχείριση των διαδρόμων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δώσει περισσότερη ουσία, περισσότερα εργαλεία στους φορείς διαχείρισης, στους διαχειριστές του δικτύου. Θέλαμε να διοριστεί ένας διευθυντής και να δοθεί ένα νομικό καθεστώς στο φορέα. Η λύση του Συμβουλίου είναι δύο επίπεδα διακυβερνήσεως. Το ένα επίπεδο είναι το κράτος μέλος με εκτελεστικό Συμβούλιο και σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου των χειριστών των δικτύων. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτή τη λύση, αλλά δεν θα πρέπει όμως να αμφισβητήσουμε ή να υπονομεύσουμε την ανεξαρτησία της ε, δράσεως των χειριστών των υποδομών. Άλλο βασικό θέμα ήταν ποια προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί στις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες. Υπάρχουν ανάμεικτα αισθήματα όσον αφορά τη δυνατότητα να δοθεί προτεραιότητα στι ε, στις εμπορικές αμαξοστοιχίες σε αυτούς τους διαδρόμους. Πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβούλια μπορεί να αποδώσει, μπορεί να επιλύσει και προβλήματα με τους επιβάτες. Εστιάζουμε τη δράση μας ε, επί κάποιων διαδρόμων, όχι επί όλου του δικτύου και προσπαθούμε να καθορίσουμε διαδικασίες για τα εμπορεύματα εκείνα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν συστήνουμε να έχει προτεραιότητα όλο ο τομέα των εμπορευμάτων αλλά τα εμπορεύματα εκείνα που χρειάζεται αξιοπιστία, ακρίβεια, χρονική όσον αφορά την παράδοση. Μέσω καλή συνεργασία των χειριστών των υποδομών θα μπορέσουμε πιστεύω να αυξήσουμε το δυναμικό των διαδρόμων, τον όγκο των εμπορευμάτων που μεταφέρεται από τους διαδρόμους και θα πρέπει να είναι και ευέλικτος ορισμός του διαδρόμου. Δηλαδή είναι ένας βασικός άξονας το, ο διάδρομος αλλά και εναλλακτικέ διαδρομές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια αυτού του άξονα. Έτσι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το δίκτυο. Το ευρωπαϊκό δίκτυο είναι πάρα πολύ εκτεταμένο, άρα υπάρχουν περιθώρια ελιγμών για να δημιουργήσουμε τους διαδρόμους αυτούς. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι η πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει ότι μέσω καλής αλληλουχίας σειρμών μπορείς να επιτύχεις βελτιστοποίηση μεταξύ Μετακίνηση εμπορικών αμαξοστοιχειών και επιβατικών αμαξοστοιχειών χωρίς να επηρεάζονται πολύ οι επιβατικές αμαξοστοιχίες. Άρα βασικό, βασική λέξη, όπως είπε και ο Σκράμερ, είναι η ευελιξία. Και νομίζω ότι η λύση που βρήκε το Συμβούλιο θα μπορούσε να αποτελέσει συμβιβασμό ακόμα και αν θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εστιαστούμε πολύ στις ανάγκες των επιβατών να έχουν προτεραιότητα, διότι αν γίνει αυτό, η πρόταση δεν θα αφορά τις εμπορικές αμαξοστοιχίες, αλλά τις επιβατικές. Εν γέννη, νομίζω ότι υπάρχει τώρα η δυνατότητα να καταλήξουμε κάπου με αυτή την πρόταση. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη μεγάλη για αυτή την πρόταση, κυρίως τώρα κατά την περίοδο της κρίσης η πρόταση αυτή θα μπορούσε να δώσει επαρκείς εγγύησεις στον πελάτη. Μπορεί να είναι σίγουρος ότι μπορεί να πάει η εμπορική αμαξοστοιχεία το σημείο Α στο σημείο Β εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και με καλές επιδόσεις όσον αφορά την ακρίβεια εκτέλεση του δρομολογιού. Αυτό θέλει ο πελάτης για να μπορεί να ανταγωνιστεί με τις οδικές μεταφορές. Αυτά έχω να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μαρινέσκου. Θέλετε να ολοκληρώσετε τη συζήτησή μας, να κλείσετε. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια και τα σχόλιά τους. Όπως είπα και στην αρχή, πιστεύω ότι τα δύο βασικά θέματα προς συζήτηση θα είναι η επιλογή των διαδρόμων καθώς και το θέμα των προτεραιοτήτων. Αναφερόμενος στο πρώτο θέμα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό που θα πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε είναι κατά πόσο η επιλογή αυτή θα γίνει μετά την θέση σε ισχύ του κανονισμού, αυτό που προτείνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή αν θα έπρεπε ευθύ εξ αρχής να γίνει η επιλογή και αν θα πρέπει να κάνουμε την επιλογή μέσω παραρτήματος, κάτι που προτείνει το Συμβούλιο. Είναι θέμα αρχής, θα πρέπει να αποφασίσουμε από αυτόν και μετά μπορούμε να συζητήσουμε εκτενώς την αρχιτεκτονική των διαδρόμων. Αυτό μπορεί να γίνει όμως μόνο από τη στιγμή που θα επιλέξουμε από τις λύσεις. Τη λύση του Συμβουλίου ή τη λύση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, κάποια από τα θέματα που εθίγησαν πιστεύω ότι καλύπτονται από το κείμενο Αναφέρομαι στα κριτήρια το πεδίο εφαρμογή. Νομίζω ότι οι ερωτήσεις που ετέθησαν βρίσκουν απάντηση στο κείμενο της ε, πρότασης. Μπορούμε να βρούμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά μας. Χαίρομαι διότι πιστεύω ότι ακούγοντας τις παρεμβάσεις των μελών ε, μου δημιουργήθηκε εντύπωση ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πολιτική συμφωνία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Υποθέτω ότι όλοι έχετε ικανοποιηθεί, ότι έχετε εσείς εντολή να προχωρήσετε ως συζητητής τις συνομιλίες με το Συμβούλιο, ούτω ώστε να καταλήξετε σε κάποια συμφωνία επί Σουηδικής Προεδρίας. Νομίζω ότι έχετε τη σύμφωνη γνώμη των μελών. Καλώς κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε πιο νωρί. Αν συντονιστέ θα ξεκινήσουν πιο νωρί, αν περιμένουμε. Ο Ντέρκ θέλει να ξεκινήσει νωρίτερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ομοφωνία. Για ναι. Θα ξεκινήσουμε τώρα, αν συμφωνείτε. Όσον αφορά τους άλλους, θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Στις 9.